Bene, Ευχαριστούμε τον Επιτροπό Ταγιάννη που ήρθε στην Επιτροπή μας, είχε μια μικρή καθυστέρηση λόγω του φόρτου εργασιών του και εμείς συχνά έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Τον ευχαριστούμε που βρίσκεται εδώ παρόν μαζί μας σήμερα. Θα προσπαθήσω να κερδίσω λίγο το χαμένο χρόνο δίνοντας το αμέσως το λόγο. Ε, ε, κύριε Γκροστέτη, θέλει να μιλήσει. Παρακαλώ, όχι. Ωραία, λοιπόν, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή Λία, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Σήμερα η μέρα ήταν πολύ έντονη και όσον αφορά τα ζητήματα που σας αφορούν. Ε, είχα μεγάλες συζητήσεις κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης ε, με τους επιτρόπους εσωτερικής αγοράς ε, που, την οποία προέδρευσε ο πρόεδρος Μπαρόσο από τις 8 και μετά τη συνεδρίαση των επιτρόπων κατά τη διάρκεια της οποίας κρίναμε ένα έγγραφο στο οποίο υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα της ανάπτυξης με επικέντρωση στην βιομηχανική πολιτική, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την πρόσβαση στις πιστώσεις και μετά είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου που μίλησε για τα, ευρωομόλογα, για τα project bonds και συζήτησε το ρόλο που θα μπορούσε να έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και στις 16 του μήνα θα λάβει χώρα μια συνεδρίαση της Επιτροπής αφιερωμένη στην ανάπτυξη για προετοιμασία της 30 ε, του μήνα όπου οι επίτροποι θα πρέπει να ε, εγκρίνουν την αναπτυξιακή πολιτική και πριν από, την από το έκτακτο συμβούλιο της 23ης. Είμαι λοιπόν πολύ ευχαριστημένος όπου όχι μόνο όσοι ασχολούνται τα μέλη του Κοινοβουλίου και οι αρμόδιοι επίτροποι του τομέα. Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε για άλλη μια φορά να δεσμευτεί ισχυρά υπέρ τη ανάπτυξη. Δεν μπορεί ωστόσο να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς μια ισχυρή δράση πολιτική, βιομηχανική πολιτική για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με όλα αυτά λοιπόν τα επιχείρηματα θα συζητήσουμε μαζί διότι κοινό μας στόχος είναι να επαναδρομολογήσουμε την ανάπτυξη με στόχο την αύξηση της απασχόλησης μέσω της προώθησης της βιομηχανικής μας βάσης. Για αυτό το σκοπό ζήτησα από τη διευθυνσή μου, τη γενική μου διεύθυνση. Όπως γνωρίζετε έχουμε νέο γενικό διευθυντή, τον κύριο Τανιέλ ε, Κρέσπο, ο οποίος πιστεύω έχει ήδη έρθει να σας συναντήσει. καθορίσαμε λοιπόν τις προτεραιότητες και την ατζέντα για τους επόμενους μήνες. Στόχος της επαναδρομολόγησης της ανάπτυξης ε, έχει ακόμη πιο κρίσιμη σημασία αν εξετάσουμε ορισμένα στοιχεία τα οποία κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Δυστυχώς η Κομισιόν προβλέπει κάμψη του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος κατά 0,3% κατά τη διάρκεια του έτους με βαθμία βελτίωση μόνο στις αρχές, στα τέλη του φετινού έτους, στις αρχές του επόμενου. Ταυτόχρονα προβλέπουμε ότι οι κύριοι δίκτυοι εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων θα καταγράψουν αισθητή επιδείνωση ένα ακόμη πιο ανησυχητικό μήνυμα φτάνει από τα στοιχεία της ανεργίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ανεργία μπορεί να φτάσει το 11% εντός της Ευρωζώνης, που είναι το χειρότερο ποσοστό από τη στιγμή εισαγωγής του ενιαίου νομίσματος. Φυσικά αποτελεί καθήκον δικό μας ε, των πολιτικών να υποστηρίξουμε με σημαντικές αποφάσεις τη ζωτικότητα των επιχειρήσεων τόσο σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργώντας τις συνθήκες για μια αηφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη. Λέγαμε στις Βρυξέλλες όπως και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όλοι εργάζονται εντατικά ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση. Κατά τις τελευταίες εβδομάδες ε, διαπίστωσα εγώ ο ίδιος προσωπικά πως ε, αυτή η ανάπτυξη αποτελεί επίγον ζήτημα τόσο για την Ιρλανδία, για την Ελλάδα, για την Ισπανία όπου συνάντησα τους πρωθυπουργούς και όπου συνάντησα επίσης ε, και την πραγματική οικονομία. Ήρθα σε επαφή με αυτήν η στόχη και οι ανησυχίες είναι ίδιες. Η οικονομία πρέπει να αρχίσει να αναπτύσσεται ξανά σε βιώσιμα επίπεδα, διαφορετικά οι πολιτικές λιτότητες που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή με τόσο θάρρος δεν θα αρκέσουν για να οδηγήσουν τις χώρες και την Ευρώπη εκτός κρίσης την ίδια εβδομάδα συνάντησε επίσης την καγκελάριο Μέρκελ και τον ε, αντικαγκελάριο Μέσλερ και η Γερμανία μου φαίνεται επίσης ότι έχει απόλυτη συνείδηση ότι η υπερβολική χρέωση, υπερχρέωση σχετίζεται επίσης με τις απόλυτες ανταγωνιστικότητες, δηλαδή τη δυνατότητα ανάπτυξης. Είναι αδύνατο να μην σκεφτούμε ε, και τα αποτελέσματα, να μην λάβουμε υπόψη και τα εκλογικά αποτελέσματα του περασμένου Σαββατοκυριακού που είχαν ε, μέσα στι άκρες, ε, έδωσαν το ίδιο μήνυμα στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα και στην Ιταλία παρότι με διαφορετικές ε, λεπτομέρειες σημείωσαν τη δυσαρέσκεια όσον αφορά ορισμένες επιλογές ή τουλάχιστον μία λάθος κατανόηση των επιλογών που έχουν γίνει. Σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο ότι οι, Ευρώπη, οι λαοί της Ευρώπης, οι συμπολίτε μας, μας ζητούν ισχυρή δράση προς υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας. Όσον αφορά εμένα, αλλά πιστεύω και όσον αφορά και την ίδια την Κομισιόν, ολόκληρη την Κομισιόν, δεν έχουμε σκοπό να αποφύγουμε αυτή την πρόκληση. Μελετάμε ήδη αυτή τη στιγμή, όπως είπα, μία σειρά από πρωτοβουλίες συμπληρωματικές που θα ενισχύσουν τις ήδη, τις ήδη επιλογές ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των πολιτών. Εγώ έχω αναλάβει μια συγκεκριμένη δέσμευση στο να καθοδηγήσω και να επιταχύνω τη μετάβαση προς μια τρίτη βιομηχανική επανάσταση στην οποία η Ευρώπη θα πρέπει να ηγηθεί. Η πρώτη επανάσταση ήταν ε, η εισαγωγή του ατμού. Η δεύτερη, εκείνη η οποία ε, εμφάνισε ένα νέο πρωταγωνιστή το πετρέλαιο και τώρα έχει έρθει η ώρα να σκεφτούμε λόγω των όσων συμβαίνουν ε, άλλες, άλλα ενδεχόμενα τα δεδομένα, τα στοιχεία μιλούν καθαρά. Κάθε χρόνο αυξάνεται ο παγκόσμιος πληθυσμός κατά 70 εκατομμύρια άτομα. Ήδη το 2030 θα έχουν διπλασιαστεί οι καταναλωτικές ανάγκες σε ενέργεια ε, ως ε, εκείνο το έτος ε, εδώ στο 2030 θα εισάγουμε στην Ευρώπη 80-90% πετρέλαιο και αέριο και θα αυξηθούν επίσης οι καταναλώσεις αγαθών, οι κατανάλωση αγαθών, ενέργειας και πρώτων υλών. Όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία και τα μέσα μεταφορά στον κόσμο το 2030 θα έχουμε 1 δισεκατομμύριο 600 εκατομμύρια οχήματα το 2050, 2,5 δισεκατομμύρια σε σχέση με τα 800 εκατομμύρια που έχουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να αναρωτηθούμε μπορούμε να συνεχίσουμε να προχωράμε με τις τεχνολογίες και τα μέσα παραγωγής που έχουμε σήμερα. Η απάντηση είναι προφανώς όχι. Τι θα βρίσκεται στο κέντρο αυτής της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης. Κατά την κρίση μου η γνώση, η καινοτομία και η αποτελεσματικότητα των πόρων που απαιτούνται για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η διαδικασία υλοποιείται ήδη. Αλλά αν δεν το συνοδεύουμε. Εάν δεν συνεχίσουμε να ακολουθούμε το δρόμο που έχουμε ξεκινήσει, θα πληρώσουμε υψηλό τίμημα όσον αφορά απώλεια ανταγωνιστικότητας, ανεργίας και διάβρωσης της βιομηχανικής βάσης της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης. Γι' αυτό θα μιλήσουμε στις 29 Μαΐου φέτος στις Βρυξέλλες στο συνέδριο Mission Growth, στο οποίο θα συμμετέχουν πολλοί ε, Ευρωπαίοι Υπουργοί Βιομηχανίας, ε, Γενικοί Διευθυντές Μεγάλων Επιχειρήσεων, η Πρόεδρος ε, της Δικής Επιτροπής Αμαλία Αρτόρη και με συντονιστή τον Τζέρεμι Ρίφκιν για τις διάφορες συζητήσεις. Στόχος αυτού του συνεδρίου θα είναι να συμβάλλει στην αναθεώρηση της νέας βιομηχανικής πολιτικής που εμείς επεξεργαζόμαστε και έχουμε την πρόθεση να παρουσιάσουμε και την οποία έχουμε την πρόθεση να παρουσιάσουμε αμέσως μετά το καλοκαίρι. Εμείς περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε νέες πηγές και η βιώσιμη ανταγωνιστικότητα είναι το business, οι επιχειρήσεις. Ε, ε, βιώσιμη ανταγωνιστικότητα σημαίνει να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την ανάπτυξη, την ενεργειακή απόδοση, την απόδοση των πόρων, μειώνοντας τα απορρίμματα και τα απόβλητα και διασφαλίζοντας την ενεργειακή ασφάλεια. Αυτά θα μας οδηγήσουν στην πολιτική μας στρατηγική και σε αυτή, θα συνοδεύεται από τη ε, θεματολογία της πρόσβασης, της πιστώσης, τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης της αγορές και τη βιομηχανική καινοτομία. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν δύο βασικοί τομείς βιομηχανικής τους οποίους θα ήθελα να σταθώ για λίγο περισσότερο. Πρώτα απ' όλα η ναυπηγική τομέας που υφίσταται τεράστια βαθιά κρίση που υπάρχει κίνδυνος να συνεχιστεί μέσα στους επόμενους μήνες. Όπως είπα, στην τελευταία μας συνάντηση έχει ξεκινήσει ένα, μια επανεξέταση της στρατηγικής leadership και έχει δημιουργηθεί μια ομάδα συντονισμού με στόχο να εγγυηθεί την επιβίωση αυτού του στρατηγικού τομέα και την ισχυρή του όθηση ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρουν αναδυόμενες αγορές, την καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες. Ελπίζω ότι η ομάδα συντονισμού θα καταφέρει μέχρι το φθινόπωρο να συντάξει μια έκθεση με συστάσει και βάσει αυτών θα προχωρήσουμε για την υιοθέτηση της νέας στρατηγικής Leadership 2020 προς τις αρχές του επόμενου έτους. Ο άλλος τομέας είναι ο τομέας των αυτοκινήτων. Η ομάδα υψηλού επίπεδου, ο 21, που ξεκίνησε το 2010, μόλις ε, είχα γίνει εγώ επιτροπό της βιομηχανίας βρίσκεται σε καλό δρόμο. Αποφασίσαμε να μετατρέψουμε την τελευταία συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου της ΚΑΡΣ 21 σε αυτή τη φάση εκκίνησης μιας νέας ε, στρατηγικής που θα πρέπει να μας δώσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την επαναδρομολόγηση και την υπεράσπιση του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Εν ώψη μάλιστα της ανακοίνωσης ε, για τα αυτοκίνητα 2020 ε, που προβλέπεται για το φθινόπωρο του 2012. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να σας ενημερώσω ότι την περασμένη εβδομάδα συνάντησα τον Λούρι Κέλμαν, Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας ε, ε, Συνδικάτων ε, των Βιομηχανιών Μετάλλων και τον Σέρτζο Μαρκέονε, πρόεδρο της ΑΤΣΕΑ ε, ένωση των ε, Αυτοκινητοβιομηχανιών ε, της Ευρώπης. Στο κέντρο των συζητήσεων μας βρίσκονταν τα μέτρα που πρέπει να συμπεριλάβουμε σε ένα σχέδιο δράσης ευρωπαϊκό για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Τρία είναι τα θέματα κλειδιά που πρέπει πιστεύω να μελετήσουμε ώστε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του τομέα των αυτοκινήτων. Πρώτο, η τεχνολογική leadership της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω της έρευνας, της καινοτομίας και της κινητοποίησης των οικονομικών πόρων που υπάρχουν διαθέσιμοι σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Έχω πρόθεση να συνεχίσω μέσα στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές ε, αυτή τη στρατηγική που εμείς υλοποιήσαμε στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Επίσης, ε, ελπίζω για καλύτερες έξυπνες ρυθμίσεις για ένα πιο απλό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει την ποιότητα και την απόδοση χωρί περιττό κόστο. Τρίτο σημείο, η υποστήριξη τη παγκοσμιοποίηση τη Ευρωπαϊκή Βιομηχανία μέσω δράσεων επικεντρωμένων στην διασφάλιση ισότιμης πρόσβαση των ευρωπαϊκών προϊόντων στους παγκόσμιε αγορές και στην πρόθεση τη εναρμόνισης των προτύπων και των τεχνικών κανονισμών. Ο κοινό παρονομαστή όλων αυτών των σενάριων είναι η καινοτομία. Ολόκληρη η οικονομία βρίσκεται υπό μετασχηματισμό αυτή τη στιγμή. Και ε, αυτή τη στιγμή βλέπετε την εμφάνιση νέων τεχνικών ε, παραγωγή που βασίζονται στι ψηφιακές τεχνολογίε, σε προηγμένα υλικά, σε βιοτεχνολογίε, σε, ε, σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, σε διαστημικέ ε, εφαρμογές, ρομποτική, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και στην επανάχρηση πρώτων υλών. Έτσι περνάμε από μια κλασική βιομηχανία σε μια νέα ε, βιομηχανία για τις μεταφορές, για τις οικοδομές, για τη χημική και την αγροβιομηχανία. Με το Horizon 2020 η Κομισιόν σκοπεύει να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. Δεν θα το συζητήσουμε σήμερα εδώ, είχαμε πολλές φορές την ευκαιρία να το συζητήσουμε, αλλά ήθελα αντιθέτως να σας παρουσιάσω ό,τι αφορά το δικό μου τομέα και τι σκοπεύουμε να κάνουμε στο μέλλον, χάρη στην υποστήριξη, στη στήριξη που ελπίζουμε να διασφαλιστεί στο επόμενο κοινό στρατηγικό πλαίσιο, ειδικότερα όσον αφορά τις ε, key ε, enabling technologies και το διάστημα και την πράσινη οικονομία, τρεις τομείς που θεωρώ ότι βρίσκονται στο κέντρο αυτής της ε, νέας βιομηχανικής επανάστασης. Ας δούμε τις ΚΕΤ, τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας χάρη στην πράσινη οικονομία και στις ε, βασικές αυτές τεχνολογίες ε, η Κομισιόν έχει ανακοινώσει ότι θα προσθέσει μια ανακοίνωση φέτος το καλοκαίρι για αυτό το ζήτημα. Τι είναι η ΚΕΤΣ. Είναι τα τεχνολογικά τουβλάκια ας πούμε με τα οποία θα οικοδομήσουμε ε, την τεχνολογική μας ανάπτυξη μέσα στα επόμενα χρόνια. φωτονική, οι νανοτεχνολογίες και οι υπόλοιπε τέτοιες τεχνολογίες έχουν τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης μια έκθεση από τους εμπειρογνώμονες της δικής μας ομάδας υψηλού επίπεδου για τους ΚΕΤΣ εκτίμησε ότι αυτός ο τομέας ήδη αξίζει σήμερα 650 δισεκατομμύρια ευρώ και θα συνεχιστεί να αυξάνεται η αξία του θα φτάσει στο 1 δισεκατομμύρια ευρώ στο 1 εκατομμύριο ευρώ εντός τριών ετών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρωταγωνιστούν σε αυτόν τον τομέα οι μεγαλύτερες, οι περισσότερες εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτό το τομέα είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι τεχνολογίες μας θυμίζουν τις αδυναμίες της Ευρώπης όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να διατεθούν στην αγορά. Γι' αυτό το λόγο εγώ πιστεύω ότι μαζί θα πρέπει να εργαστούμε ώστε η έρευνα να εφαρμόζεται όλο και περισσότερο στη βιομηχανία. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που θα μπορούσε να ενδιαφέρει αυτή την Επιτροπή αφορά τις πρώτες ύλες. Όπως γνωρίζετε έχουμε ξεκινήσει αυτή την εταιρική σχέση για την καινοτομία των ε, πρώτων υλών, για την αντικατάσταση και για την ανακύκλωση. Τους επόμενους μήνες θα βρεθώ και στη Γρελανδία για να υπογράψω μια νέα σύμβαση για τις πρώτες ύλες μέσα στις επόμενες ε, μέρες και μήνες ε, θα πάω και στην Κολομβία και στις Ηνωμένε Πολιτείες για να ε, ασχοληθούμε με αυτό το θέμα που είναι στρατηγικά σημαντικό. Ο εισηγητή τη σχετική έκθεση για το Κοινοβούλιο γνωρίζει πολύ πόσο σημαντικό είναι ένα άλλο θέμα, είναι αυτό τη διαστημική πολιτική. Έχουμε εργαστεί εντατικά σε αυτό το τομέα μια νομοθετική πρωτοβουλία ανακοίνωση για το θέμα της ε, επιτήρησης και της επιχειρησιακής ε, γνώσης στο διαστημικό τομέα που θα αφορά τις δραστηριότητες επιτήρησης και παρακολούθησης των διαστημικών αντικειμένων επιτήρηση και μετρολογικές προβλέψεις και παρατήρηση των αστεροειδών και των μετεωρητών θα συνεχίσουν όπως προηγουμένως όσον αφορά το Γαλιλαίο εγώ αντιλαμβάνομαι ότι πλατιάζω λίγο, αλλά είναι μεγάλος ο τομέας μου, πολύ ευρύς ο τομέας που ασχολούμαι και περιλαμβάνει μια σειρά από θέματα για τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να ενημερωθεί αυτό το Κοινοβούλιο. Σας επιβεβαιώνω ότι 28 Σεπτεμβρίου θα λάβει η χώρα το δεύτερο μεγάλο γεγονός ε, συμβαντού Γαλιλαίου θα ε, στείλουμε στο διάστημα δύο ακόμη δορυφόρους και ήδη από το 2014 θα ξεκινήσουμε να ενεργοποιούμε υπηρεσίες και θα φτάσουμε στον πλήρη αστερισμό το 2018. Αστερισμό δορυφόρων φυσικά. Ε, εσείς γνωρίζετε ποιο είναι το θέμα που αφορά το έγνος. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το έγνος μεταξύ Συμβουλίου, Κομισιών για την προϋπολογισμό και για τη χρηματοδότηση της το GMS GNS είναι ένα θέμα που μας προβληματίζει επειδή η Κομισιόν προτείνει ε, πέραν των ε, να έχουμε πέραν των ε, προϋπολογισμών και των χρηματοδοτήσεων του GNSS μπορεί να φαίνεται αντίφαση αλλά τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να ζητάνε από την Κομισιόν χωρίς να αυξηθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός να πράξει κάτι ή αυξάνεται ο κοινότικό προπολογισμό, ή ε, διαφορετικά εμείς δυσκολευόμαστε να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μας ζητάνε για το GMS. Δεδομένων όλων αυτών, ε, εμεί έχουμε χρηματοδοτήσει μέχρι του πρώτου μήνε του 2014 και θα κάνουμε ό,τι μας είναι δυνατόν ώστε να, ε, να γίνει εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου το 2014 πρόθεσή μου ήταν να σας παρουσιάσω την αναθεώραση ε, του REACH όπως έχει προβλεφθεί μέχρι τον Ιούνιο. Σήμερα αξιολογούμε την εμπειρία κατά τα πρώτα χρόνια υλοποίηση του κανονισμού χάρη στι εκθέσεις από τα κράτη-μέλη το 2010 και από τον οργανισμό το 2012. Σε αυτό το πλαίσιο η Κομισιόν έχει την πρόθεση να ε, υπερβεί τους απλά νομικούς, τις απλά νομικές υποχρεώσεις και να συμπεριλάβει στην αναθεώρηση αξιολογήσεις του κόστους των διοικητικών ε, δαπανών και της επίπτωσης στην κοινοτομία. Τελευταίο θέμα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πρόσβαση σε πιστώσεις. θα ήθελα να ζητήσω την βοήθεια του Κοινοβουλίου. Καθώς συζητάμε για τις μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές, κυρίως όσον αφορά το πρόγραμμα COSME, το οποίο αφορά πέρα από την καινοτομία και την έρευνα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προβλέπει, πρωτο, προβλέπει πρωτοβουλίες ε, για την παγκοσμιοποίηση, δράσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας για μας, Όλο αυτό είναι εξαιρετικά σπουδαίο. σπουδαίο. Ένα άλλο θέμα για το οποίο θα ήθελα να σε ενημερώσω είναι ότι την περασμένη Τετάρτη μαζί με τον Επιτροπό Μπανιέ στείλαμε μια επιστολή στον Ανδρέα ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής για να ζητήσουμε η εφαρμογή της Βασιλείας 3 να μην έχει επιπτώσεις κακές, ε, άσχημες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ζητήσαμε αναθεώρηση της εφαρμογής των κανονισμών, των κανόνων του Βασιλεία 3 ώστε το ποσοστό επικινδυνότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βασιστεί, να χαμηλώσει από το 75% στο 50%. Φυσικά, αφού αναγνωριστεί αυτή η μικρότερη επικινδυνότητα, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να υποφεληθούν από αυτό, ανεξάρτητα από το αν είναι πελάτες ε, τραπεζών με τυποποιημένο έλεγχο ή με εσωτερικό έλεγχο, διότι για την καινοτομία και την ανάπτυξη είναι βασικό να μπορεί να υπολογίζει κανεί του απαραίτητου χρηματοδοτικού πόρου. Και όταν είναι κανεί μικρό, το να λάβει πίστοση δεν είναι εύκολο. Η έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από 10 μέρες περίπου, μας το επιβεβαιώνει επιπλέον. Σας ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας. Προσπάθησα να είμαι εξαντλητικός και να σας τα παρουσιάσω όλα. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά όπως βλέπετε είναι πολλά τα θέματα με τα οποία απασχολούμαστε μαζί για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μια ισχυρή αναπτυξιακή πολιτική και να δώσουμε απαντήσεις στους Ευρωπαίους πολίτες. Μάλιστα ευχαριστούμε τον Επίτροπο που μας δημιούργησε όμως ένα πρόβλημα όπως γνωρίζουμε όλοι. Δηλαδή είναι 3 και 45, στις 4 η ώρα έχει προβλεφθεί η ψηφοφορία. Οπότε είχαμε προβλέψει τη συζήτηση από τις 3 ε, μέχρι τις 4 μόνο. Ε, Έχω 12 εγγεγραμμένους και καταρχήν θα ήθελα να πω ότι κλείνω την, ε, τον κατάλογο των υποψηφίων για να λάβουν τον λόγο, 13 όχι 12. Μπορείτε απλούστατα να κάνετε μία σύντομη ερώτηση για να υπάρξει και απάντηση. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να μας επαρκέσει ο, ο χρόνος. Έχουμε ένα τέταρτο το πολύ. Γι' αυτό σε ένα τέταρτο μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι θα υπάρξει ψηφοφορία. Λοιπόν, ε, μία ερώτηση ο καθένας ενός λεπτού και προχωράμε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σε ένα λεπτό η ερώτησή μου. Θα επικεντρωθώ σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι ένα από τα θέματα που συζητάμε αυτή την εποχή και κεντρικό και για την Επιτροπή μας. Ορίζοντας 2020 και τα προγράμματα που το συνοδεύουν, όπως το COSME, που επιτρέπει ένα οικοσύστημα προκειμένου μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν περισσότερες διευκολύνσεις ώστε να αναπτύξουν τις πρωτοβουλίες τους και άρα την ανάπτυξη. Σχετικά με αυτό το πρόγραμμα λοιπόν έχω να σας ρωτήσω το εξή. Όπως γνωρίζετε κύριε Επίτροπε, το προηγούμενο κόσμο, το chip όπως το λέγαμε, γιατί βέβαια δεν είναι ακριβώς το ίδιο, περιλάμβανε συγκεκριμένες δράσεις όπως το προήμνο, όπως το Ευρώπη Καινοτομία, τη χρηματοδότηση, την εφαρμογή που στο κόσμο δεν αναφέρονται. Όλα αυτά τα στοιχεία δεν αναφέρονται στο κόσμο. Λέτε ότι αργότερα θα συμπεριληφθούν με λεπτομέρειες στο καθετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, παρόλο που δεν έχουμε τις λεπτομέρειες τώρα και θα τις έχουμε αργότερα, 2014 κτλ. Μήπως θα μπορούσατε να μας αναφέρετε κάποιες δράσεις για τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί αυτή η δράση κόσμε. Ο επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο και δεν χρειάζεται να περιοριστεί κανείς την ενέργεια. Προηγουμένως θέλω να σας ευχαριστήσω ευχαριστήσω ότι αναφερθήκατε εις ε, τις εκλογές στη Γαλλία και χαίρομαι ιδιαίτερο γιατί και η καγκελάριος μας επανεκάλυψε την ανάπτυξη στην Ευρώπη και θα είναι προς καλός όλων. Χρειάζεται μια νέα στρατηγική αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη όπως ε, είπατε. Ξέρετε ότι η κατάσταση είναι δυσχερής. Πώς είναι δυνατόν δυνατόν το Κοινοβούλιο να έχει ε, δυνατότητες στο στη διαδικασία αυτή διότι κατά τη γνώμη μου δεν ε, ακολουθούν όλη ε, την πολιτική που έχει αποφασιστεί οπότε πρέπει να δούμε τι γίνεται στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρέπει να δούμε τι γίνεται στο επίπεδο της ΕΣΑ, αν θα προχωρήσουμε δηλαδή στο πρόγραμμα αυτό ή όχι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις για τον Επίτροπο. Έγινε μία μελέτη το 2009 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είδαμε ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντικές ε, οι μελέτες για να μπορεί κανείς να ενημερωθεί για την κατάσταση στον τομέα της τεχνολογίας. Ακόμη όμως υπάρχει δυσκολία όσον αφορά την πρόσβαση ε, στις προδιαγραφές διότι ακόμη εκπονούμε προδιαγραφές αντί να τις εφαρμόζουμε. Θα ήθελα λοιπόν αν μέσα στα πλαίσια του πρόγραμμα COSME η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξασφαλίζει πρόσβαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα αυτό. Επίσης όσον αφορά το ενιαίο δίπλωμα ευρασιτεχνίας. Ε, πολλοί έχουν κατακρίνει ότι η τωρινή ε, μορφή είναι εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οπότε πρέπει να δούμε ε, στον ε, τομέα της τεχνολογίας εάν υπάρχουν προβλήματα. Ευχαριστώ. Ε, Έχω λάβει από την περιοχή μου πολλά παράπονα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις για καθυστερήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν, όταν απευθύνονται ε, και δεν αναφέρονται τα θέματα αυτά εις την ατζέντα του 2020. Οπότε τι μέτρα λαμβάνετε και για την τεκμηρίωση και για την την ατελή κατανομή των πόρων, τη σύγχυση για το ποιος ε, ευθύνεται γιατί και σε ποιον πρέπει να απευθυνθεί κάποιος για να ε, διατυπώσει παράπονα. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επιλύσει τα προβλήματα αυτά σε επίπεδο προγραμμάτων. Οπότε τι κάνετε, ο κύριος Έλμερ. Κυρία η Πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω τον Επίτροπο εάν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μία πανικόβλητη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις πρόσφατες εκλογές στη Γαλλία και στην Ελλάδα και αν υπάρχει ε, μία συνεκτική απάντηση. Λέτε ότι πρέπει να αυξήσουμε τον προπολογισμό αλλά η Ευρώπη δεν έχει χρήματα, έχει μόνο χρέη. Οπότε ε, πρέπει πρέπει να αντιληφθείτε τους λόγους για την απώλεια ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης που οφείλεται σε υψηλή φορολόγηση. Δεν χρειαζόμαστε έξυπνες ρυθμίσεις αλλά λιγότερες ρυθμίσεις και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ε, όσο πρέπει να γνωρίζουμε ότι όσο η Ελλάδα και η ε, Πορτογαλία παραμένουν στον ευρώ ποτέ δεν θα ξαναγίνουν ανταγωνιστικές και για την κλιματολογική πολιτική λέτε ότι η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί της ε, τρίτης βιομηχανικής επαναστάσεως αλλά αντιτίθε, αντιτάσσεται η Αμερική με το πετρέλαιο από σχιστόλιθο ή η Ινδία και η Κίνα με νέες τεχνολογίες και θα ήθελα να μου πείτε εσείς τι κάνετε για να λύσετε τα προβλήματα που υπάρχουν. Ευχαριστώ κύριος Ράνσντορφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορείτε να Μπορείτε να περιγράψετε τα συγκεκριμένα μέτρα που θα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιταχύνει την τρίτη βιομηχανική επανάσταση. Ευχαριστώ, Γκρόστετ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, η η ε, ανάπτυξη δεν είναι κάτι το οποίο διατάσουμε και ε, ε, διεπίστωσε ότι στην προεκλογική εκστρατεία δεν μιλήσαμε αρκετά για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας και βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις μας είναι καταχρεωμένες και εδώ συμφωνώ κύριε Επίτροπε ότι οι μόνες που μπορούν να δημιουργήσουν πλούτο και θέσεις εργασίας που χρειαζόμαστε είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάζεται όμως περισσότερη ευελιξία, λιγότερη ρύθμιση και χρηματοδότηση, την οποία να αναφέρεται. Ε, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει δημιουργία κεφαλαίων κινδύνων ευρωπαϊκών ε, και ε, βοήθεια και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα έπρεπε να υπάρξει δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα συμμετέχουν μεγάλοι επενδυτές που θέλουν να προωθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τη Γρυλανδία μπορείτε να μας ενημερώσετε διότι η Κίνα είναι σε αντιπαράθεση με την Ευρώπη και ανταγωνίζεται για την πρόσβαση στις σπάνιες γέες, οπότε θα, να μου πείτε τι γίνεται. Ο κύριος Τσουκαλάς. Ευχαριστώ κύριε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για το ζήτημα που θίξατε σχετικά με τα μέτρα που σκέφτεται να πάρει η Κομισιόν σε συνδυασμό με τα εκλογικά αποτελέσματα σε Γαλλία και Ελλάδα. Ελπίζω να γίνει κατανοητό ότι σε όσες χώρες δοκιμάζονται από την κρίση γίνουν εκλογές, τα ίδια αποτελέσματα θα παίρνατε σαν και αυτά της Ελλάδας. Και τούτο διότι τα μέτρα αυστηρότητος χωρίς συνδυασμένη ανάπτυξη δεν οδηγούν πουθενά. Θα ήθελα λοιπόν κύριε Επίτροπε να συνεχίσετε την προσπάθειά σας αυτήν που λέτε ότι αρχίσατε στην Κομισιόν έτσι ώστε ένα νέο μοντέλο ε, αυστηροποίησης των δημόσιων οικονομικών μαζί με προσπάθειες ανάπτυξης να φέρει ευτυχέστερα αποτελέσματα και να σκεφτόσαστε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι τα αίτια αλλά τα αποτελέσματα μιας πολιτικής. Ευχαριστώ, Ρόι. Σαν Επίτροπε, είμαι μεταξύ των πολιτικών που πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει δράση και όχι υπερβολικά προγράμματα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι έγινε μία ανακοίνωση πρόσφατα για την βιομηχανική πολιτική. Σε όλα τα νομοθετικά μέτρα στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει να δούμε κατά πόσον επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας Οπότε θα μπορέσει δηλαδή να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία και να μην παραμείνει στα χαρτιά. Ευχαριστώ κύριε Σκόμιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ ότι ε, ε, ε, με κάθε θυσία πρέπει να εξοικονομήσουμε, αλλά αυτό δεν επαρκεί. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι επαρκεί η εξοικονόμηση, δεν έχουμε, ε, ε, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ε, το πρόγραμμα COSME είναι περιορισμένο. Τι άλλες δυνατότητες λοιπόν μπορούν να υπάρξουν για διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μια καλή πρόταση είχε ε, διατυπωθεί στο Νέο Δελχή για μια πλατφόρμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την αντιφάνισή τους στην αγορά. Η κυρία Μέρκης. Ε, σας ευχαριστώ διότι όντως η ανάπτυξη είναι το πιο σημαντικό και πρέπει να έχουμε μία πολιτική κινήτρων αλλά τα κίνητρα χρειάζονται και συγκεκριμένα μέτρα. Πολλά ακούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο αλλά δεν βλέπουμε συγκεκριμένες ενέργειες. Οπότε πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν ε, να γίνουν συμφωνίες ε, για πρώτες ύλε, αλλά τι περιμένετε σαν αποτέλεσμα από τη στρατηγική για τις πρώτες ύλε. Και πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ζωτικές και πρέπει να δούμε εάν θέλετε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα τι επιπλέον μπορεί να προσφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να είναι καινοτόμες ή να έχουν προϊόντα υψηλής ποιότητος πράγμα το οποίο δεν είναι προφανές. Και τέλος όσον αφορά την νανοτεχνολογία πιστεύω ότι και ο τομέας αυτός χρειάζεται ανακαίνιση. Τι μπορούμε να προσβλέπουμε στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βεμπέρ. Ευχαριστώ. Το πρώτο θέμα. Με ναι, ακούτε, δεν με ακούτε είναι το εξή. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις αποτελούν θύματα της, ε, το θέμα του ανταγωνισμού. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να απευθυνθούν ε, στο, στην υπηρεσία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτές. Τι σκοπεύετε να κάνετε κύριε Επίτροπε προκειμένου να διευκολύνετε την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα όργανα αυτά έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον αθέμητο ανταγωνισμό. Τις επιδοτήσεις δηλαδή που δίνονται ε, αθέμητα στους ανταγωνιστές τους. Οι δημόσιες αγορές σε πολλές χώρες μας είναι κλειστές. Η κινέζικη αγορά, για παράδειγμα, είναι κλειστή στις χώρες μας. Του Καναδά, επίσης, σε ένα μεγάλο βαθμό. γιατί ο Μποβαρδίε μπορεί να βάζει στο Παρίσι τις ράγες ε, τρένων η ε, μετρό, εμείς όμως δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο στον Καναδά. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό. Ευχαριστώ, ο κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Την περασμένη εβδομάδα ήμουνα στα Ηνωμένα Εμμυράτα όπου υπάρχει μία νέα ζώνη ελευθέρου εμπορίου χωρίς φορολογία είτε κεφαλαίου είτε εταιριών και υπάρχουν ήδη 30.000 απασχολούμενοι. Θα ήταν δυνατόν κύριε Επίτροπε η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων να κοιτάζει πώς μπορεί να καταργήσουμε έναν χάρτη πορείας ε, για τις επιχειρήσεις και τη φορολογία τους ε, μέχρι το 2020 για να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε μια ευκαιρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να το αφήνουμε ε, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας μόνο το έργο αυτό. Θα πρέπει να εμπλακεί και η Γενική Διεύθυνση Enterprise κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχουν μόνο οι πιστώσεις αλλά να δούμε τι μέλη γενέστε παρακάτω παρακάτω. Ε, κύριε Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις προς εσάς. Γνωρίζω την ε, τεράστια προσπάθεια που κάνετε υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ε, μάλιστα με αρκετή πρωτοτυπία γιατί δημιουργήσατε ένα χώρο για να βοηθάτε τις καινοτόμες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα ψηφιακά, κάτι πολύ βασικό <clears throat> για την Ευρώπη. Διαπιστώνω ότι κάθε φορά όμως υπάρχει ως ενδιάμεσος κάποια εθνική αρχή. Και εκεί γίνεται η στρέβλωση, γιατί βλέπετε ότι οι, πάνε στους διαγωνισμούς δεν πάνε επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι που είναι διάμεση τα ίδια κερδίζουν. Οπότε γνωρίζετε εσείς, μπορείτε να μου πείτε πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτήν την μόνιμη παρουσία των ενδιάμεσων ε, παραγόντων του κράτους. Έπειτα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει δυνατότητα να προβάλλουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μερικές φορές οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, ζητούν από τις μικρές να τις βοηθήσουν στην καινοτομία, αλλά αυτές οι μικρές δεν εμφανίζονται πουθενά, είναι αόρατες. Άρα χάνουν την αγορά θα ήταν δυνατόν να υποχρεώσετε όταν οι μεγάλες ε, οι επιχειρήσεις ε, δίνουν υπεργολαβία στις μικρές επιχειρήσεις για την καινοτομία να μπορεί ε, να μπορούν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις να είναι παρούσες και να φαίνονται, να προβάλλονται για τη δουλειά που κάνουν. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τι ερωτήσει. Δίνουμε πέντε λεπτά στον Επίτροπο για να συνεχίσουμε με την ψηφοφορία. Προετοιμαζόμαστε στο μεταξύ για την ψηφοφορία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλε τι ερωτήσει. Θα ξεκινήσω απαντώντα στην ερώτηση στην οποία υπογραμμίστηκε το πώς έχει κάνει λίγα η Κομισιόν για την Ανάπτυξη και ότι ξύπνησε μόλις πρόσφατα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι για ανάπτυξη εγώ μιλάω, δεν ξέρω αν με ακούτε, Κατηγορήσατε λοιπόν την Κομισιόν ότι ασχολήθηκε θα ήθελα να υπενθυμίσω στον ε, αξιότιμο κύριο Έλμερ ότι από την αρχή της εντολής της θητείας μου μίλησα για την ανάπτυξη και συνάντησα στη Μεγάλη Βρετανία, στη χώρα σας, στη συντηρητική κυβέρνηση μελετώντας προσεκτικά τα έγγραφα της αναπτυξιακής πολιτικής της συντηρητικής κυβέρνησης ε, πριν από πέντε εβδομάδε μίλησα με τον Δούκα του Ιόρκ και τον ε, αρμόδιο υπουργό για τη διαστημική τεχνολογία τη Βρετανία. Μιλήσαμε για αναπτυξιακή πολιτική, για τη σπουδαιότητα του διαστηματο και για τα όσα ε, λαμβάνει υπόψη η Βρετανική κυβέρνηση και η Βρετανική βασιλική οικογένεια για το διάστημα. Θα οργανώσουμε στο Λονδίνο μια σημαντική εκδήλωση το Σεπτέμβριο για την εκτόξευση των πυράβλων του Γαλιλαίου και το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες Γαλιλαίου υπέρ της ανάπτυξης. Ε, όσον αφορά το ερώτημα και πάλι παραμένουμε στο διάστημα, ε, εγώ έχω την πρόθεση να προχωρήσω μπροστά σε όλα τα μέτωπα. Το πρόβλημα είναι ότι στο Συμβούλιο το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το πρόγραμμα GMES. Η, η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών ζητάει οι χρηματοδοτήσει του GMES να περιλαμβάνονται στον κοινοτικό προπολογισμό. Μόνο η Πολωνία και η Λιθουανία είναι υπέρ της πρόταση της Κομισιόν να έχουμε χρηματοδότηση του GMS e εκτός του κοινοτικού προϋπολογισμού. Εγώ πιστεύω ότι το σημαντικό είναι να προχωρήσουμε και μετά θα βρούμε μία λύση για να χρηματοδοτήσουμε ένα έργο εξαιρετικής σπουδαιότητας για την ε, γεωπαρατήρηση, για την καταπολέμηση της κλιματικής αναλλαγής, αλλά και για την παγκοσμιοποίηση του επιχειρηματικού μας συστήματος ε, ουσιαστικά στην Αφρική, στην Ασία και σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Όσον αφορά τώρα την καθυστέρηση των ε, πληρωμών εκ μέρους της Κομισιόν, ο αξιότιμος κύριος Φόρντ έχει δίκιο. Εμείς ε, κάνουμε, δίνουμε μάχη για να λαμβάνουν τα κράτη-μέλη όσα λάμβαναν προηγουμένως η οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές ε, και αν υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου καθυστέρησε η Κομισιόν λόγω διαφορών υποχρεώσεων να μου το γνωρίσετε διότι εάν ε, μπορώ θα επέμβω αμέσως. Το γραφείο μου είναι στη διάθεσή σας και αν Δεν ξέρω αν η μετάφραση γίνεται σωστά. Εγώ αυτό είπα. Εάν υπάρχουν περιπτώσεις να μου τις επισημάνετε και εγώ θα παρέμβω αμέσως ώστε να τις, επιλύσω. you, I... Συζητώ μαζί σας. Είμαι έτοιμος για να βρούμε μια καλή λύση. Αγαπητή κυρία, ε, εάν υπάρχουν προβλήματα θα κάνω ό,τι μπορώ για να βρούμε μια ικανοποιητική λύση με τη Γενική μου Διεύθυνση. Όσον αφορά το πρόγραμμα COSME, εμείς έχουμε μόνο 2,5 δισεκατομμύρια στην πρόταση προϋπολογισμού μας. Μπορούμε να συμπεριλαβούμε και άλλα πράγματα και τα επιχειρηματικά κεφάλαια, τα venture capital που όπως ε, υπογραμμίστηκε εδώ τα venture capital έχουν ήδη προβλεφθεί, έχουμε ήδη θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τα venture capital. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ακόμη περισσότερες διασφαλίσεις, θα δημιουργήσουμε Ήδη με το παλιό σύστημα, με το τρέχον πρόγραμμα ΣΥΠ, καταφέραμε να χρηματοδοτήσουμε 146.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση στα κεφάλαια. Εμείς θα θέλαμε να προχωρήσουμε. Το φαινόμενο μόχλευσης που μπορούμε να διασφαλίσουμε, το leverage με το πακέτο COSME, θα ε, συνοψιστεί στη διάθεση 25 δισεκατομμυρίων. Στη συζήτηση για το κόσμο ίσως μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ουσιαστικά όσον αφορά τις ε, συγκεκριμένες ε, δράσεις για τις key enabling technologies και για τις πρώτες ύλες, όσον αφορά τις πρώτες ύλες, Έχουμε μια innovation partnership η οποία αποφασίστηκε και ξεκινάει αυτή τη στιγμή για την αντικατάσταση και την ανακύκλωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει φυσικά να συμμετέχει. Για πιο συγκεκριμένα τώρα Πιο συγκεκριμένα τώρα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε σκοπό μέχρι το 2020 για την ανακύκλωση και την αντικατάσταση. Θέλουμε να ξεκινήσουμε 10 ε, καινοτόμε δράσεις πιλωτικές τουλάχιστον για τις θεμελιώδεις εφαρμογές, να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της χρήση των υλικών, να αναπτύξουμε την έρευνα και να επεξεργαστούμε στατιστικά εργαλεία ευρωπαϊκά με ένα σύστημα υποδειγμάτων, μοντέλων και εφαρμόζοντας μια προενεργό στρατηγική πολυμερή. Όσον αφορά τον ορισμό των ανοηλικών, στις 28 Οκτωβρίου 2011 η Κομισιόν υιοθέτησε, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο, μια σύσταση για τον ορισμό των ανοηλικών και αυτή τη στιγμή η Κομισιόν εργάζεται ώστε να μπορέσει να διευκρινίσει τα τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την ερμηνεία των ανοηλικών, ώστε να ε, καθιερώσει έναν τρόπο μέτρησης. Ε, γίνονται αυτή τη στιγμή διαβουλές μεταξύ των υπηρεσιών όσον αφορά την παραποίηση. Το μελετάμε, αποτελεί δέσμευση προτεραιότητα τη Κομισιόν. Ξέρετε πόσο έχουμε μαχηθεί και εμεί μαζί με το Κοινοβούλιο για το ζήτημα του. Οι λύσει δεν είναι εύκολε. Ε, έχουμε αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια στο Συμβούλιο όσον αφορά την αμοιβαιότητα, όπως γνωρίζετε εσείς μαζί με τον Επίτροπο Μπαρνιέ έχουμε ε, συντάξει μια επιστολή προς τον Πρόεδρο Μπαρόζο για να θέσουμε το πρόβλημα της ε, υπεράσπισης ε, ε, εμείς θέλουμε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό ο οποίος να επαληθεύει τις δράσεις που σχετίζονται με έξω ευρωπαϊκές επενδύσεις όπως αυτή που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, πριν από τέσσερις εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Επιτρόπη υιοθέτησε για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ανέφερε ο κ. Βέμπερ, μια πρόταση υπόψη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που σχετίζεται με το θέμα της αμοιβαιότητας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Η πρόταση φέρει την υπογραφή των Επιτρόπων Μπαρνιέ και Γούχτα που την οποία εγώ υποστηρίζω και επί του ουσία. Όσον αφορά το τελευταίο που ήθελα να πω, θέλω να απαντήσω όσον αφορά την εφαρμογή της βιομηχανικής πολιτικής. Εμείς ε, υλοποιούμε αυτή τη στιγμή όλες τις δοκιμές ανταγωνιστικότητας. Το competitiveness proofing έγινε δεκτό με μεγάλο θυσιασμό από πολλές χώρες τις οποίες εγώ έγραψα ώστε να υιοθετηθούν αμέσως. Γνωρίζετε ότι υπήρξε ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο οποίο παρουσιάστηκε μία ε, φωτογραφία της Ευρώπης ε, με φως και ε, σκιά. Στη Γερμανία η πρόταση έγινε δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό από τον κύριο Ρέσλερ ο οποίος σκοπεύει να υποστηρίξει τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το competitiveness proofing. Για όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις παραμένω στη διάθεσή σας και για μια ενδεχόμενη μελλοντική συνάντηση. Ελπίζω ότι σε κάθε περίπτωση το γραφείο μου, η γενική μου διεύθυνση θα βρίσκονται στη διάθεσή σα, στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να σα παρέχουν όποιε πληροφορίε ετηθείτε. Και πάντα χαίρομαι να συναντώ τα μέλη του Κοινοβουλίου εδώ και 15 χρόνια. Για 15 χρόνια υπήρξε ε, βουλευτή σε αυτό εδώ το Κοινοβούλιο και τώρα βρίσκομαι στην άλλη πλευρά του Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, εκ μέρους όλης της Επιτροπής ζητάμε συγγνώμη για το τα κάναμε τα πράγματα λίγο γρήγορα για τη σύγχυση, αλλά όπως ξέρετε έτσι γίνεται πριν από τις ψηφοφορίες, χρειάστηκε να βιαστούμε. Ευχαριστούμε για την ε, πολυπλήρη σας ολοκληρωμένη έκθεση και για τις απαντήσεις σας και θα σας ξαναδούμε σύντομα. Ευχαριστούμε, καλή δουλειά. Bene, Ας ξεκινήσουμε αμέσως τις ψηφοφορίες. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση Κάλφιν. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μία δοκιμή για να δούμε εάν έχουμε τους σωστούς αριθμούς. Είστε υπέρ και της ε, αναβολής της καθυστερήσεως με την οποία ξεκινούμε την ε, ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Θα ψηφίσω ε, διαχειρός. Κατά τα άλλα όλοι οι άλλοι συμφωνούν. Ε, είμαστε αρκετά καλά, άρα ξεκινάμε με την έκθεση Καλφίν ε, τροπολογία της ΛΥΜΠΕ 14. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Οι 15 και οι 16 είναι μαζί, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται Λίμπε 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 και 18 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Τροπολογία 19 πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Λίμπε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 και 32 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος σχετικά με την τροπολογία 33 ξεκινά ένας ΕΛΚ ε, παραπάνω από ό,τι δικαιούται εγώ δεν έχω ψηφίσει εδώ. Αποτέλεσμα. Λίγη ψηφοφορία. 11 υπέρ 45 κατά, άρα απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά,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 απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 και 59 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62-63 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 ηλεκτρονική ψηφοφορία για συνολική ψήφιση. Ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δύο ΕΛΚ πλεονάζοντες. Εγώ ήδη έβγαλα τη δική μου κάρτα, ένας ακόμη. Τώρα ένας ε, είναι πλεονάζον. Λοιπόν, λίγοι. 50 υπέρ, 7 κατά. 51, 51 υπέρ και 7 κατά. Ε, εγκρίθηκε και συγχαίρουμε τον εισηγητή. Περνάμε στη δεύτερη ψηφοφορία που αναφέρεται στην έκθεση Edith Herzog. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά έλεγχος θέλετε για ποιο ποια τροπολογία θέλετε να ελέγξουμε τη 45 μάλιστα ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινά η ψηφοφορία. Λίγη. 35 υπέρ, 24 κατά, άρα εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 50 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Λίγη ψηφοφορία. Ε, ένα σοσιαλιστής πλεονάζων. Λίγοι, 31 υπέρ, 28 κατά. 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά,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 κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος για την 84. Λίγη. Ένα ΣΕΛΚ πλεονάζει. 32 υπέρ, 27 κατά. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει εγκριθεί αλλά ας κάνουμε έναν έλεγχο γιατί δεν είμαι πολύ βέβαιη ελέγχουμε την 90 την 90 τροπολογία 90 λίγη ο ηλεκτρονικός έλεγχος 41 υπέρ 18-19 κατά εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 8, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, απορρίπτεται, με συγχωρείτε, 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 172 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 176 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 180 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές να το ελέγξουμε. έλεγχος της τροπολογίας 8 ψήφισαν όλοι κλείνει η ψηφοφορία 41 υπέρ 18 κατά ήταν πολύ σαφές αλλά δεν το είδα εγκρίνεται λοιπόν τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε. Τροπολογία 11. Ελέγχουμε. Κλείνει η ψηφοφορία. 29 προς 29. Αλλά έχουμε και μία ψηφοκατά. Α, υπέρ. 30 προς 29 εγκρίνεται. Τροπολογία 11 ήταν αυτή. Τροπολογία 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32, υπέρ 32 τροπολογία τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ίντα 1 υπέρ κατά μου φαίνεται ότι απορρίπτεται αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά το chiuso. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Είναι τα, ένα. Είναι τα δύο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 Αφετ 4 υπέρ κατά αποχή. Όλες τις αφετ μαζικά. Συμφωνείτε όλοι. Όλες οι τροπολογίες αφετ μαζί από την 4 έως την 14. Συμφωνείτε. Ωραία λοιπόν από 4 έως 14 υπέρ κατά Κύριε Τσίτσεστερ, κατά μαζικά ή θέλετε να ψηφίσετε μία προς μία. Ε, κυρία Πρόεδρε, ήμουν υπέρ του να ψηφίσουμε μαζικά από την 4 μέχρι τη 10. Γιατί πιστεύω ότι αλλιώ υπήρχε ένα κενό. Ε, από την 4 έως τη 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Από, αφετ 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά,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 48 υπέρ, 11 κατά, μία αποχή, συγχαρητήρια, η γνωμοδότηση, η έκθεση έχει εγκριθεί. Ας περάσουμε στον εισηγητή κύριο Χατζηγεωργίου. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 13 τροπολογία, 16 ε, τροπολογία συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 17 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 17. Ελέγχουμε την 17. Κλείνει η ψηφοφορία. 31 υπέρ, 29 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 Ελέγχουμε τη συμβιβαστική 2. Ηλεκτρονικά πρώτα. Ελέγχουμε τη συμβιβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. 20 υπέρ 39 κατά. Συνεπώς απορρίπτεται η συμβιβαστική 2. Τροπολογία 19. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ελέγχουμε την 25 Κλείνει η ψηφοφορία. 32 προς 28 εγκρίνεται ή 25 ωραία 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ελέγχουμε την 27 περίεργη αυτή η ψηφοφορία λέει η πρόεδρος. Ε, η πλειοψηφία είναι περίεργη. Ε, κλείνει η ψηφοφορία. 29 υπέρ, 31 κατά, απορρίπτεται. Η 28 τώρα. Υπέρ, κατά, η λίστη ψηφίζεται, απορρίπτεται. Τουλάχιστον οι επικεφαλής αντιπροσωπείων πρέπει να όταν πρέπει να ψηφίζουν προς την αυτή αλλιώς δεν καταλαβαίνει 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές ας κάνουμε έναν έλεγχο ας κάνουμε έναν έλεγχο ηλεκτρονικό 31 τροπολογία κλείνει η ψηφοφορία εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 37 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται, λέει. Ας κάνουμε τον έλεγχο. Λοιπόν, για την 37. Τροπολογία 37. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά οι πλειοψηφίες ε, ε, δεν είναι σταθερές. Ε, αλλάζουν σε κάθε ψηφοφορία. Κλείνει ψηφοφορία 19 υπέρ, 37 κατά. Απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ με την τροπολογία την προφορική υπέρ, 10 ε, συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω για την τροπολογία 5 ελέγχουμε ηλεκτρονικά Κλείνει η ψηφοφορία. 16 υπέρ, 43 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία ένα ΕΛΚ επιπλέον. «51 υπέρ, 52 υπέρ, 3 κατά, 4 αποχές, εγκρίνεται συγχαρητήρια». Περνάμε στην έκθεση Σιμάνσκι, συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. συμβιβαστική, Τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 3, 6 ε, συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για την 8 να ψηφίσουμε. Ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 8. Τρόπολ κλείνει ψηφοφορία. 28 υπέρ, 29 υπέρ, 30 κατά. Απορρίπτεται. Είχα δίκιο όμως, οι πλειοψηφίες είναι πολύ κοντινές ε, τελικά.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 επιλύθηκε το πρόβλημα του ε, παραπάνω έλκα η 57 υπέρ ένας κατά μια αποχή εγκρίνεται συγχαρητήρια περνάμε στην έκθεση Ζούμπερ τροπολογία 19 με προφορική τροπολογία παρακαλώ Συνάδελφα Μέρκης, θέλατε να πείτε κάτι. Πρόεδρε, ευχαριστώ που το αναφέρατε, διότι υπάρχει μια προφορική τροπολογία που προτείνετε λόγω κάποιας νομικής διατύπωσης. Αν θέλετε, μπορώ να σας διαβάσω το κείμενο, αλλά νομίζω ότι το έχετε όλοι, πιθανώ στην λίστα ψηφοφορία σας. Ευχαριστούμε. Δεν θέλει κανείς να διαβάσουμε το κείμενο. Όχι. Παίρνουμε λοιπόν τροπολογία 19 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 ε, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, ε, εγκρίνεται συγγνώμη 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές 25 δεν είμαι σίγουρη ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά τροπολογία 25 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 25, τροπολογία 25 απορρίπτεται τροπολογία 10 υπέρ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 αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά να ελέγξουμε πια την 46 Κλείνει η ψηφοφορία 31 υπέρ 27 κατά εγκρίνεται Ζητώ συγγνώμη, 47 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές μου φαίνεται ότι έχει εγκριθεί, ωστόσο μπορούμε να το ελέγξουμε. Κλείνει. 32. κατά. Απορρίπτεται λοιπόν 24 θετικής ψήφοι. Αυτό ισχύει για το 14, λοιπόν 15 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 10, 2 μάλλον. Τροπολογία 2 υπέρ κατά, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία, τελ, ε, συγγνώμη, τελική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, 55 υπέρ, μία ψήφος κατά, μηδέν αποχές. Ε, συγχαρητήρια, ολοκληρώσαμε και σήμερα γρήγορα την ψηφοφορία και περνάμε τώρα στην έκθεση. του κυρίου Κανσιάν για τα καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το λόγο, δώστε ένα λεπτό ώστε να, βγούμε, να βγουν όσοι βγουν από την αίθουσα. Ας αφήσουμε ένα λεπτό ώστε να αναχωρήσουν όσοι είναι να αναχωρήσουν. E- λοιπόν, όσοι δεν έχουν κάποιο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, ας αναχωρήσουν. Παρακαλώ. Bene. Allora, iniziamo, proseguiamo. Συνεχίσουμε λοιπόν τις εργασίες μας δίνοντας τον λόγο στον κύριο Καντσιάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θεωρώ ότι το σημερινό θέμα, παρότι εδώ μιλάμε μόνο για μια γνωμοδότηση, θα πρέπει να έχει τη δέσμευσή μας δεδομένου ότι πρόκειται για το θέμα της εποχής αφού μιλάμε πολύ για προγραμματισμό. Στη συνέχεια θα πρέπει να βρούμε όμως και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και τις αντιστοιχείς δυνατότητες για να μπορέσουμε να επενδύσουμε στις υποδομές και να τις υλοποιήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η γνωμοδότηση βασίζεται σε τρία σημεία κλειδιά για την υποστήριξη της ανάπτυξης, γιατί όλοι Όλο μιλάμε για ανάπτυξη. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταλάβουμε κιόλα ε, που θα την βρούμε και πώς πρέπει να πράξουμε. Εγώ διακρίνω τρία σημεία κλειδιά. Σε αυτή τη γνωμοδότηση το πρώτο σημείο είναι ο εξορθολογισμός και ο συντονισμός. Υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά μέσα, πολλά προγράμματα χρηματοδότησης διαφορετικά, τα οποία συχνά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε αυτή την πολυμορφία δημιουργείται και σύγχυση και αβεβαιότητα μεταξύ των όσων θέλουν να την αξιοποιήσουν τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Κατά την άποψή μου λοιπόν χρειάζεται ένα καθαρό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει όλα τα μέσα και τη σχέση μεταξύ τους. Μια ιδιαίτερη περίπτωση πιστεύω μάλιστα εμβληματική, χαρακτηριστική για να καταλάβουμε τη σύγχυση που υπάρχει είναι ότι αν δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο έλαβε μία θα έλεγα ε, σημαντική μορφή το πολιτικό πνεύμα αποσκοπούσε στο να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε πόρους ε, όχι ως χορηγήσεις αλλά ως ε, επενδύσεις με απόδοση μέσω διαφόρων νομικών γνωμοδοτήσεων διαπιστώνεται κατά την υλοποίηση ότι αυτό το ταμείο δεν μπορεί να συνάδει με τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Δηλαδή κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που είχαμε προκαθορίσει εμείς. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που μας λέει ότι πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να αλλάξουμε τη φιλοσοφία των ε, χρηματοοικονομικών μας μέσων, το να δορίζουμε χρήματα μεσοχορηγήσεων χορηγήσεων πρέπει να σταματήσει διότι πρέπει να εγκρίνουμε και να προωθήσουμε προγράμματα σωστά, υλοποιήσιμα, αποδοτικά διότι η εκκίνηση είναι δύσκολη. Εκεί πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, όχι να δορίζει χρήματα σε προγράμματα που δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους ε, υπό ένα πνεύμα οικονομικής ε, και περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Το δεύτερο σημείο είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο Επίτροπο Σταγιάννη επέστησε την προσοχή μας στου κανόνες της Βασιλείας 3 που επιτρέπουν ε, μεγαλύτερο διάστημα χρονικό για την εφαρμογή του ποσοστού επικινδυνότητας. Θεωρώ ότι οι νέες δημοσιονομικές προεπτικές ε, μας καλούν να προσέχουμε ιδιαίτερα ώστε να μην σκοτώσουμε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ όλοι εμείς δεν σταματάμε να συζητάμε για την στήριξή τους και μετά κάνουμε τα αντίθετα. Ωραίο πράγμα η χρηματοδότηση του κόσμου και το Horizon 2020 και πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να αξιοποιήσουμε όλες τις πρωτοβουλίες υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι τόσο σημαντικές για την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανακαμψή της. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε προσεκτικά τις δυνατότητες ε, αύξησης του μέγιστου προβλεπόμενου κατοφλίου της Long Guarantee Facility στο πλαίσιο του ίδιου του κόσμου. Το τρίτο σημαντικό σημείο που για μένα είναι θεμελιώδη σημασία ε, για την καινοτομία και μάλιστα ρηξικέλευθο σημείο. Όταν μιλάμε για νέα χρηματοδοτικά μέσα. Η βάση των χρημάτων είναι πάντα η ίδια. Υπάρχει κάποιος που θέλει να τα ξοδέψει αμέσως και θέλει να τα λάβουν δωρεάν τα διάφορα προγράμματα όπως το παρελθόν με τους ελάχιστους πόρους που έχουμε. Άλλοι θα θέλανε να τα μετατοπίσουν για να δώσουν κίνητρα και να πολλαπλασιαστούν μέσω διασφαλίσεων, ωστόσο μιλάμε για, πάντα για τα ίδια χρήματα. Δεν είναι ότι αυξάνονται αυτά τα χρήματα. Εδώ λοιπόν προκύπτει το τρίτο σημαντικό σημείο. Εμείς εγκρίνουμε αυτή τη στιγμή τα project bonds, τα ομόλογα προγραμμάτων όσον αφορά το κομμάτι των ε, αναπτυξιακών εταιριών που μπορούν να μπουν σε χρηματοπιστωτικές ε, αγορές και να εκδώσουν ομόλογα που θα έχουν τη διασφάλιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, εδώ μιλάμε για, ένα μια ορθή μετάβαση που θα μπορούσε να βελτιώσει ορισμένες καταστάσεις. Αλλά δεν είναι αυτή αυτό η σημαντική πτυχή γιατί αυτοί που πρέπει να μπουν στις χρηματαγορές είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μέσων της η ίδια να εκδώσει ομόλογα για την υλοποίηση των υποδομών. Διαβάζω στις εφημερίδες αυτές τις ημέρες ότι και ο ίδιος ο Μπαρόσο λέει ότι ένα σχέδιο Μάρσαλ για τις νέες υποδομές Βλέπω το αναπτυξιακό σχέδιο που αφορά τη Γαλλία με τον κύριο Λάντ που λέει στο πρώτο σημείο ότι project bond για την υλοποίηση υποδομών απευθείας με ομόλογα τα οποία θα εκδίδει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι δύο σπόρους. Αυτά αποτελούν μηνύματα τα οποία εγώ βλέπω με θετικό μάτι. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να τα κατανοήσουμε και επίσης να βλέπουμε και το χρόνο που περνάει γιατί όσο εμείς μιλάμε ε, καίγεται το σπίτι απ' έξω και ε, η κατάσταση είναι δραματική. Θεωρώ ότι τα μηνύματα τα έχουμε λάβει αυτές τις μέρες από αυτές τις ε, τελευταίες ώρες. Ε, καθήκον μας είναι λοιπόν να είμαστε θαραλέοι και να έχουμε τη βούληση να προχωρήσουμε και να πράξουμε έτσι ώστε τέλος αυτή η Ευρώπη εκτός από τη λιτότητα να σημειώσει και ανάπτυξη και να μπορέσει να αφιερώσει τις δυνατότητες και τη βούλησή της ώστε να βγει στις αγορές απευθείας και να ε, αναπτύξει όλα αυτά, να τραβήξει μαζί της όλα αυτά τα χρηματοδοτικά ε, προγράμματα να βασιστεί σε επενδύσεις μακροπρόθεσμες και όχι μικροπρόθεσμες ή μεσοπρόθεσμες, επενδύσεις για σημαντικά έργα, προγράμματα τα οποία έχουν απόδοση. Και όχι μόνο χορηγήσει που δορίζει η μεσοπρόθεσμε, να πρόκειται για επενδύσεις που θα οδηγήσουν ε, σε μια συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε χωρίς όλα αυτά, διότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια στενοπό και πρέπει όλοι να δεσμευτούμε ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το ποιοτικό άλμα. Εγώ προερχόμενος από την Επιτροπή Μεταφορών και βλέποντας τα θέματα των υποδομών, κάθε φορά τέλειος προγραμματισμός, ωραία ε, θεωρία, ωστόσο πρακτική δεν βλέπω πουθενά, διότι πάντα προσκρούμε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν χρήματα για την υλοποίηση. Αν δούμε τις περιφέρειες, τα κράτη-μέλη μας, δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ και δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να προχωρήσει κανείς ε, με κανένα παραπάνω ευρώ χρέο. Πιστεύω ότι η Ευρώπη σε αυτό το σημείο είναι ο μόνος θεσμός που θα μπορεί να και ε, έχει την υποχρέωση να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Αυτή την έκκληση κάνω προς του συναδέλφους μου για να σας πω ότι κοιτάξτε η ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί διαφορετικά παρά μόνο με αυτούς τους πόρους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Καντσάν. Το λόγο έχει ο Βιτόριο Πρόντι. Μιλώ εξ ονόματος του συναδέλφου Πίτερ Σκένερ ο οποίος δεν είναι παρόν και ζητάει συγγνώμη. Ο Πίτερ θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κύριο Καντζάν για τις προσπάθειές του για αυτή τη γνωμοδότηση. Θα ήθελε να ζητήσει συγγνώμη που δεν κατάφερε να βρεθεί εδώ σήμερα για να συμμετάσχει σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ο Πίτερ μου ζήτησε να σας παρουσιάσω μερικές από τις προκαταρκτικές του παρατηρήσεις σχέση με το σχέδιο γνωμοδότησης. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελε να διερευνηθούν διαφορετικές στρατηγικές για τα χρηματοδοτικά μέσα εν ώψη του Horizon 2020 και του COSME. Η χρηματοδότηση προγραμμάτων για τις επιστήμες και την τεχνολογία αποτελεί το θεμόλιο για να τονώσουμε την καινοτομία στην Ευρώπη μέσα στα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι πόροι θα αξιοποιηθούν στο μέγιστο. Ο Πίτερ θα ήθελε επίσης να επισημάνει τη σπουδαιότητα τη χρηματοδότηση όχι μόνο βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη, αλλά και των μακροπρόθεσμων επενδυτικών δομών, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά τα προγράμματα θα είναι βιώσιμα. Ο Πίτερ ε, γκρίνει τα συμπεράσματα του κυρίου Καντσάν στη ε, γνωμοδότησή του και προσδοκεί να συνεργαστεί με τον εισηγητή και τους κοιόδης ε, μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ζητήσω τον λόγο και για δικό μου λογαριασμό στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να ζητήσει τον λόγο. Εφόσον δεν υπάρχει κανείς, ο κύριος Καντσάν ή ο κύριος Πρόντι. Ναι, ναι, ε, από ό,τι κατάλαβα νόμιζα ότι είχατε τελειώσει. Είχα τελειώσει για λογαριασμό του κυρίου Σκίνερ και ζήτησα το λόγο και προσωπικά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για, που μου δίνετε το λόγο. Απλούστατα ήθελα να τονίσω όπως το έκανε και ο συνάδελφος Καντσάν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε σύντομα σε αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα και θέλω να τονίσω τη σημασία για τις ε, ε, διαστημικές υποδομές διότι ε, όλα τα θέματα που έχουν προταθεί είναι ε, αποδεδειγμένα ευρωπαϊκά επιτεύγματα και ε, υπάρχει μία μετατόπιση χρονική όσον αφορά το χρόνο που θα εκτελεστούν τα, ε, οι δαπάνες και με τη στιγμή που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν οι διαστημικοί σταθμοί. Γι' αυτό και πρέπει να ε, ασχοληθούμε με το θέμα αυτό διότι η υποδομή και η κατάρτισή της δεν δεν ιστερεί ε, μόνο διότι δεν εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές και θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και να μπορέσουμε να εκτελέσουμε χωρίς να χάνουμε χρόνο αυτές τις επενδύσεις διότι είναι και συγκυριακή η αξία και πολύ σημαντική των εγχειρημάτων αυτών διότι ε, πρέπει στο γενικότερο ευρωπαϊκό βιομηχανικό σύστημα να δοθούν αυτά τα κίνητρα που θα μπορέσουν να παρασύρουν και άλλες δραστηριότητες εξού και είναι απολύτως απαραίτητο τα θέματα αυτά να εκτελεστούν και να εφαρμοστούν και ιδίως εδώ αναφέρομαι εις ε, την ανεξήγητη απόφαση ε, που, του να ξεκινάμε το σύστημα GMS ε, σχετικά με την κατάρτιση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Δεν ξέρω το GMS, ο Γαλιλαίο, όλα αυτά πώς θα μπορέσουν να υλοποιηθούν και είναι θέματα τα οποία μπορούν να μας θέσουν ε, στο προσκήνιο και ε, για μερικά χρόνια με τα μέτρα που παίρνουμε ε, καθυστερούμε την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας και έχω μία σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς το Συμβούλιο διότι θα πρέπει το Συμβούλιο να κατανοήσει ότι αυτές είναι ευρωπαϊκές υποδομές και η προστιθέμενη αξία και η ανάγκη εκτελέσεώς τους κατ' εμέ είναι αδιαφυσβήτητη και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τον κύριο λόγο έχει κύριο Σοντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αισθάνομαι πολύ περίεργα στη συγκεκριμένη αυτή η φάση, γιατί δεν μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω σφαιρικά τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης απέναντι στην κατάσταση ανταγωνισμού στην οποία βρισκόμαστε με την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία κτλ. που έχουν μαζικά προγράμματα επενδύσεων στο δικό τους το, την επικράτεια. Μας λείπει λοιπόν ένα μεγάλο σχέδιο επενδύσεων για τις υποδομές Αυτά που προτείνει η Επιτροπή βρίσκονται έτη φωτός πίσω από τις ανάγκες μας. Για τις μεταφορές είχαμε υπολογίσει 600 δισεκατομμύρια ευρώ ότι χρειαζόμαστε. Σήμερα για να διατηρηθεί η πυρός μας, η Ευρώπη, σε κατάσταση ανταγωνιστική, χωρίς τίποτα περίεργο, χρειαζόμαστε περίπου 1.000 με 1.500 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2020 και πολλοί από εμά είπαμε στο Παρόζο όταν το έγραφο 2020 εμφανίστηκε, είπαμε ότι χρειάζεται ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο. Μιλάμε εδώ για καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, δηλαδή τα έσοδα που ήδη υπάρχουν. Εγώ έχω να κάνω διάφορες προτάσεις. Πρώτον, το πρώτο ευρώ που κερδίζουμε είναι αυτό που δεν θα ξοδέψουμε. Εδώ θα έλεγα να κάνουμε έναν έλεγχο των δημοσίων δαπανών σε τρία επίπεδα. Περιφέρειες, χώρες, Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας εχθρός. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει συντονισμός. Σε ολόκληρο τον πλανήτη γίνονται διπλωματικά ε, έχουμε διπλωματικά γραφεία χωρίς ούτε καν ένα φωτοτυπικό μηχάνημα. Συνεπώς, χρειαζόμαστε οικονομίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες μέλη και οι περιφέρειες. Να γίνει αυτός ο ανεξάρτητος έλεγχος, να τον κάνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο με τα 27 εθνικά ελεγκτικά συνέδρια για να δούμε όλοι μαζί τι μπορούμε να εξοικονομήσουμε χωρίς να πληγεί φυσικά η κυριαρχία κανενός είναι δισεκατομμύρια ευρώ που μπορούμε να κερδίσουμε και να τα δώσουμε στη συνέχεια για επενδύσεις. Τώρα για την καινοτόμο χρηματοδότηση. Προτείνω να κάνουμε μία σύγκριση. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Ας δούμε λοιπόν τα κράτη-μέλη πώς χρηματοδοτούν τις ανάγκες τους σε υποδομές. Είτε πρόκειται για ηλεκτροδότηση, είτε για νερό, για φυσικό αέριο. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, έχουμε χρηματοδοτήσει την Ήπεθρο, στην Ήπεθρο την ηλεκτροδότηση με ένα πολύ μικρό φόρο που δεν το κατάλαβαν καν οι καταναλωτές. Ε, παίρνουμε δηλαδή τα χρήματα αυτά από την κατανάλωση που γίνεται στη, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Μιλάμε για υποδομές και δεν ξέρουμε καν που ανήκουν οι υποδομές αυτές. Ανήκουν στους ε, παραδοσιακούς παρόχους, τηλέφωνο, ηλεκτρικό δηλαδή και φυσικό αέριο. Τελικά δεν ξέρουμε ποιος θα επενδύσει και πώς. Γιατί να μην έχουμε ένα μικρό φόρο κατανάλωσης για όλη την κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα μας διασφαλίσει τη χρηματοδότηση των υποδομών αυτών, ώστε η επικράτειά μας και οι πολίτες της να μπορούν να εξυπηρετούνται. Ο ανταγωνισμός δεν μας επιτρέπει έπειτα να χρηματοδοτούμε τους αυτοκινητόδρομους που είναι λιματικοί από εκείνους οποίοι είναι πλειονασματικοί. Είναι τρελό. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους εμπειρογνώμονές της να μας παρουσιάσει σφαιρικά πώς έχουν τα πράγματα με τα κράτη-μέλη για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ένα μεγάλο ε, σχέδιο υποδομών και επενδύσεων αναγκαίων είναι αναγκαίες. Ο Φραν Σολόντ έδωσε ένα παράδειγμα στη Γαλλία. Εντάξει, βέβαια τι έκανε, δεν ανακάλυψε τίποτα καινούριο. Έχει αντιγράψει όλα όσα έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μεγάλα σχέδια υποδομών. με πάση περιπτώσει. Πρέπει να έχουμε μια σφαιρική άποψη για τον 21ο αιώνα αν κάνουμε λάθη ή αν κάναμε λάθη, ας τα δούμε. Αυτό πάντως που προτείνεται με την ανακοίνωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν με ικανοποιεί. Έχουμε το 2020, εκεί είναι ε, συνολική η προσέγγιση. Αλλά όσον αφορά την χρηματοδότηση και τον τρόπο χρηματοδότησης, εγώ πιστεύω ότι μένει ακόμα να γίνει η δουλειά για την παρουσίαση, γιατί αυτό που έχουμε δεν είναι ικανοποιητικό. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω ότι καταρχήν ε, ο συνάδελφος έχει ετοιμάσει μια εξαίρετη έκθεση. Πιστεύω ότι λίγες διορθώσεις και διευκρινήσεις θα μπορούσαμε μόνο να κάνουμε. Για παράδειγμα λέμε ότι η Ευρώπη παλεύει για την καινοτομία. Θα πρέπει εδώ όμως να προσθέσουμε ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να κάνουμε ορθολογικές δαπάνες. Οι επιχειρηματίες επιστήνουν την προσοχή μας στο γεγονός ότι συχνά οι νομικές λύσεις δεν είναι αποτελεσματικές. Καλό θα ήταν να έχουμε πιο σφαιρικές λύσεις, οι οποίες να μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε τα κονδύλια χωρίς αυτά να κατακαιρματίζονται στα διάφορα προγράμματα. Σήμερα το πρωί είχαμε συζήτηση με εκπροσώπους των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τι μας είπαν, είπαν ότι φυσικά και πρέπει να ελέγχουμε τα κονδύλια, αλλά δεν θα πρέπει ο έλεγχος αυτός να φτάνει σε γελιότητες, να στέλνουμε επιστολές για έξοδο 20 σαντίμ, να είμαστε ορθολογιστές, να αποφεύγουμε την ανοησία. Είδαμε επίσης ότι χρειάζονται εγγύησει ώστε μακροχρόνια να διασφαλίζονται κονδύλια για την καινοτομία. Γιατί η καινοτομία δεν έρχεται με παραγγελία μέσα σε λίγο καιρό. Χρειάζονται επενδύσει προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτόμε ιδέε και λύσει. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι προτάσεις που γίνονται επιστημονικά στέκουν, ότι είναι εφαρμόσιμε. Να εξοικονομήσουμε πόρους, όπω λένε οι συνάδελφοι, αλλά να υπάρχει ορθολογισμός στις δαπάνες και επαλήθευσή τους και έλεγχό τους, αλλά με φύη τρόπο. Ευχαριστούμε. Κυρία Νίμπλερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Καντσάν για την εξαιρετική έκθεσή του. Πιστεύω ότι ανέφερε στη γνωμοδότησή του όλα τα βασικά θέματα και υπάρχουν βέβαια ορισμένα που μπορούν ακόμη να βελτιωθούν, αλλά γενικώ θεώρησα ότι η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και γι' αυτό και ήθελα να παρέμβω. Έχουμε μεγάλη ανάγκη επενδύσεων στην Ευρώπη και δεν υπάρχει αναγκαία υποδομή για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει επ' αυτού την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Είτε μιλάμε για τις οδικές μεταφορές, είτε για τις σιδηροδρομικές, είτε για το ευρυζωνικό σύστημα. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα όπου πρέπει να καταρτιστεί καλύτερα η υποδομή μας και να υπάρξει μία ευρωπαϊκή μονάδα. Συμφωνώ με τον κύριο Ομπί ότι θα έπρεπε να έχουμε μια πιο σφαιρική αντιμετώπιση και αυτό είναι δύσκολο για την Ευρώπη διότι ο κύριος Οντί ε, είπε ότι ε, δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ε, με μικρό κόστος στην Ευρώπη διότι δεν υπάρχει μια ενιαία φορολογική αρχή έχουμε χρεωμένους προϋπολογισμούς είτε ε, ανεπαρκείς προϋπολογισμούς άρα πρέπει να βρούμε εναλλακτικές πηγές χρηματοδοτήσεως να μπορούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα με εγγυήσει που θα καταρτίζεται από την έκτη αλλιώς που θα διαθέτουν ιδιωτικά κεφάλαια και θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις υποδομές. Για μένα το κρίσιμο θέμα είναι να δούμε πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ένα ιδιωτικό κεφάλαιο που θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε για επενδύσεις και ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε πιο συγκεκριμένα τις περιπτώσεις και να δούμε ε, τι είναι τα μέτρα τα οποία χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτή την υποδομή. Ευχαριστώ τον κύριο Καντσάν και έχω να πω μία φράση ακόμη στον κύριο Πρόντι. Συμφωνώ κύριε Πρόντι ότι η ώρα ε, ε, των ευκαιριών δεν πρέπει να την ε, εγκαταλείψουμε για το GMS, για το Γαλιλαίο και ότι θα πρέπει να υπάρχει μία χρηματοδότηση στα πλαίσια του κοινοτικού προϋπολογισμού και ε, γι' αυτό πρέπει ε, να μην σκεφτόμαστε μόνο το αποτέλεσμα αλλά πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε ρεαλιστικές δυνατότητες να καταρτήσουμε κάτι στην Ευρώπη, ε, Ο υπόλοιπος κόσμος δεν κοιμάται, προχωρά και πρέπει και εμείς να μπορέσουμε να μην κάνουμε τόσες οικονομίες σε αυτό το τομέα και να εξοικονομήσουμε κάπου αλλού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καντσάν. Πολύ ενδιαφέρον που... Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούγαμε και την Κομισιόν, αλλά δεν είναι εδώ. Αρκετές από τις ερωτήσεις ε, ήταν για την Κομισιόν. Καλό θα ήταν λοιπόν να ήταν εδώ θα μου άρεσε επίσης, να... ήθελα επίσης να μάθω ότι σκέφτεται για όλα αυτά οι Κομισιόν. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι η συζήτηση μεταξύ των λίγων που βρίσκονται εδώ, όσα άκουσα με ικανοποίησαν ιδιαίτερα όλοι οι ομιλητέ. Θεωρώ ότι όλοι αναφέρθηκαν στα πραγματικά επίγοντα θέματα. Αναφέρομαι στο κύριο Ντόδη ε, ειδικότερα που ανέφερε έναν ε, ε, πολιτικά επιχειρήματα τα οποία συμμερίζομαι μίλησε για τον εξορθολογισμό του τεραστίου σχεδίου υποδομών για τις επενδύσεις και για το μέλλον πιστεύω ότι αν θεωρήσουμε ότι η χρηματοδοτική πόροι, τα 40 συν 10 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής αρκούν για να μπορέσουμε να τραβήξουμε, να φέρουμε εις πέρας ε, σε σύντομο χρονικό διάστημα την συλλοποίηση που θέλουμε για την ανταγωνιστικότητα. Θεωρώ ότι είμαστε εκτός του δρόμου που θα θέλαμε να ακολουθήσουμε. Εάν θεωρήσουμε ότι κάποιος άλλος, κάποιο κράτος μέλος ή κάποια περιφέρεια θα μπορέσει να τα καταφέρει έτσι, κάνουμε λάθος. Το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι αυτές οι υποδομές που εμείς προγραμματίζουμε, που εμείς αποφασίζουμε να υλοποιήσουμε, θα παραμείνουν ε, μέσα στα έγγραφά μας. Αυτό είναι που με αποθαρρύνει. Είναι σαφές ότι αν καταφέρουμε να παρέμβουμε με εξορθολογισμό των υπαρχών των κονδυλίων θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε κάποια ουσιαστικά κονδύλια. Αλλά πόσο χρόνο έχουμε για να πράξουμε κάτι τέτοιο, πώς θα το πράξουμε. Σε δέκα χρόνια ίσως θα πετύχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω αντιθέτως ότι η διαγωνιστικότητα και η οικονομία σήμερα μας φωνάζουν μας καλούν να κάνουμε κάτι αμέσως. Αύριο πρωί πρέπει να κινητοποιήσουμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες για την υλοποίηση αυτών των μεγάλων έργων. Τις προάλλες μαζί με τον συναδελφό Νίμπλη ήμασταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όταν μιλάμε για ευρυζωνικό δίκτυο που εδώ μιλάμε για 20 MB, εκεί φτάνουν τα 300, τα 120 MB και εξυπηρετούν το 80% των χρηστών. Μιλάμε για νούμερα που εμείς δεν έχουμε καν ονειρευτεί στην Ευρώπη. Ούτε καν τα έχουμε ονειρευτεί. Εγώ όταν ακούω τέτοιες ταχύτητες, ότι στον κόσμο υπάρχει κάτι τέτοιο που μας ξεπερνάει σε όλα τα θέματα. Ο, ο, ο κόσμος αρχίζει και μα ξεπερνάει στα πάντα εκτό από, από την ηλικία και από τα θέματα τη γύρανσή. Είμαστε μια λίγο ηλικιωμένη Ευρώπη, αυτό είναι ένα άλλο θέμα φυσικά. Αλλά θεωρώ ότι πραγματικά πρέπει να συνταχθούμε όλοι μαζί ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Οι διαστημικέ υποδομέ. κύριε Πρόντι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σα, ε, με τον Γαλιλαίο και την GMES που σχετίζονται μεταξύ τους στενά θα έπρεπε να προχωρούν μαζί. Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε κομμάτι κομμάτι το Γαλιλαίο και να ξεχνάμε το GMS e επειδή έτσι δεν θα καταφέρουμε ποτέ να υλοποιήσουμε πραγματικά ε, τις επενδύσεις μας. Ε, έχει... Θα χρειαζόμασταν και συμμετοχή δημοσίου και ιδιωτικού ε, τομέα επίσης ε, σε αυτό το τομέα έχουμε και όλα τα θέματα των μεταφορών, των ενέργειας, ε, των επικοινωνιών, όπως έλεγα προηγουμένως, κατά την άποψή μου. Έναν πολύ απλό υπολογισμό, με στοιχεία από εδώ και από εκεί από την Κομισιόν, μιλάμε για 1150 δισεκατομμύρια ευρώ για τα διάφορα έργα. Για να απαντήσω στη συνάδελφο Νίμπλε και να πω πώς θα μπορέσουμε να έχουμε τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Εάν εγώ θεωρώ ότι ένα χρηματοδοτικό έργο, για οποιαδήποτε υποδομή σήμερα δεν ολοκληρώνεται ποτέ στο 100% με την πρώτη χώριση που δίνουμε σε μια τέτοια αναπτυξιακή εταιρεία με δημόσια επέμβαση 30% εμείς θα τραβήξουμε και τον ιδιωτικό τομέα στην επένδυση. Αυτή είναι η πρόκληση αν είχαμε λοιπόν τα 500 δισεκατομμύρια από τα 1150 θα τραβούσαμε όλους τους υπόλοιπους ε, στα προσελκύαμε όλους τους υπόλοιπους σε αυτή την υλοποίηση. Αυτό θα είναι το ποιοτικό άλμα που εμείς θα πρέπει να επιτύχουμε μέσω των σχεδίων, θα έλεγα, εξορθολογισμού, αλλά και μέσω των σχεδίων ανάπτυξης ε, για το εγγύς μέλλον μας. Συμφωνώ απόλυτα. Με το... Μιλάμε για τα τρία επίπεδα. Βρισκόμαστε σε μια δραματική κατάσταση σήμερα. Χρειαζόμαστε να έχουμε ένα συγκεκριμένο ε, τραπέζι για τις περιφέρειες, ένα για τα κράτη-μέλη και μια άλλη συνεδρίαση για την Ευρώπη, ώστε να μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις και να δούμε τι μπορούμε να εξοικονομήσουμε από τις δαπάνες ποιον παράγοντα θα μειώσουμε και ποιον θα αυξήσουμε, ποιον παρονομαστεί. Συνεπώς καλό είναι να υπολογίζουμε και να ε, μεριμνούμε για τις δαπάνε, αλλά δεν πρέπει να επιμένουμε σε αυτή την ύφεση. Και αυτό θα γίνει μέσω, κατά τις αποψή μου, αυτού του συστήματος και μέσω αυτής της σημαντικής δοκιμής ε, την οποία έχει να αντιμετωπίσει δοκιμασίες που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί ε, και μάλιστα γρήγορα. Και σταματήσουμε να μιλάμε με ολολόγια για την ανάπτυξη όταν με ανάπτυξη εννοούμε την φυσιολογική ανάπτυξη, τη δημιουργία της ε, ενιαίας αγοράς που θα μπορούσαν να είναι οι φυσιολογικές δραστηριότητες μιας ανάπτυξης που έχει μια χρονική συνέχεια. Πρέπει να κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα. Και αυτό το άλμα χρειάζεται θάρρος για να γίνει. Ευχαριστώ κύριε Καντσάν. Σας υπενθυμίζω ότι η ημερομηνία προθεσμία για τις τροπολογίες είναι Τετάρτη 23 Μαρτίου 12 το μεσημέρι, ε, Μαΐου, συγγνώμη, 12 μεσημέρι και ότι ψηφοφορία στην ΙΤΡΕ 19 Ιουνίου ε, στην budget 20 Ιουλίου και στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο του 2012 φέτος. Όσον αφορά τις λοιπές πληροφορίες που πρέπει να σας δώσω είναι τις 29 Μαΐου από τις 3 έως τις 4.30 θα έχουμε μία κοινή ακρόαση Ήτρε και Ρέτζι για το Horizon 2020 και την περιφερειακή πολιτική. Και ότι ως Επιτροπή θα συνεδριάσουμε 30 και 31 Μαΐου πρωί και απόγευμα και τις δύο μέρες ε, από τις 9 έως τις 18 και 30. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας και καλό βράδυ.